We still have to discuss one item on our... Έχουμε και άλλο θέμα σήμερα σε διάταξη. Uh, the report on Iran. Έκθεση για το Ιράν. Προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ιράν. Σας παρακαλώ, ας αρχίσουμε. The rapporteur is Mr. Belder. Εισηγητής είναι ο κύριος Belder. He's there, so uh... Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα να αρχίσουμε. Παρακαλώ κύριε Βέλντερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να περιμένω για να μιλήσουμε. Έχουμε διάφορα πηγαδάκια εδώ, μήπως ενοχλώ. Thank you very much. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε, λέει ο Μπέλντερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα του Ιράν εδώ και καιρό απασχολεί το Κοινοβούλιο. Πιο πρόσφατα απεφάθη το Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμα το Φεβρουάριο φέτος στο Στρασβούργο. Το ψήφισμα αυτό μπορεί να αποτελέσει καλή βάση για την εργασία στην Επιτροπή μας για μια έκθεση ε, σχετικά με τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιράν. Από την άλλη, το πολιτικό τοπίο έξι μήνες αργότερα έχει κάπως αλλάξει. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εγκρίνει νέες κυρώσεις γιατί το Ιράν ε, συνεχίζει μάλλον εφόσον συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Πάντω η κατάσταση παραμένει ζωφερή και η πολιτική κατάσταση στο Ιράν. Στο ψήφισμα αυτό η Επιτροπή μας έχει την ευκαιρία τώρα να ενημερώσει την πολιτική της για το Ιράν, να τη διευρύνει ταυτόχρονα και να την εμβαθύνει. Σε συνεργασία με όλους τους συναδέλφους προσβλέπω να κάνουμε καλή δουλειά και θα έχει τέσσερα κεφάλαια το σχέδιο έκθεσης μου. Πρώτον, εσωτερική πολιτική κατάσταση στη χώρα. Ε, θέματα ε, όπως η κατάσταση της αντιπολίτευσης, ε, ο επίμονος κατασταλτικός χαρακτήρας κυβέρνηση απέναντι στον πληθυσμό, η έλλειψη διαδικασίας εκδημοκρατισμού στη χώρα και η κατάσταση της οικονομίας χώρας ε, μεταξύ ε, αυτών και εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα. Κεφάλαιο δεύτερο, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Συλλαμβάνονται διαδηλωτές και μέλη της αντιπολίτευσης αυθαίρετα, αλλά και το θέμα της μεταχείρισης των κρατουμένων είναι πολύ σημαντικό. Και με πρωτοβουλία κάποιων συναδέλφων τονίζουμε και θέματα ελευθεροτυπίας, ε, και εδώ μιλώ για έντυπο τύπο αλλά και για ηλεκτρονικό ε, ψηφιακό. Αυτό που με ενδιαφέρει επίσης είναι η συμπεριφορά απέναντι σε εθνικές και θρησκευτικέ μειονότητες και θα δώσω έμφαση στην ε, έκθεσή μου. Τρίτο κεφάλαιο, εξωτερικές σχέσεις του Ιράν. Θα ήθελα εδώ λίγο να μιλήσω για τις σχέσεις με την Τουρκία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία και τις υπόλοιπες χώρες του Περσικού κόλπου. Οι σχέσεις του Ιράν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Ρωσία επίσης θα μας απασχολήσουν. Και ένα τελευταίο κράτος που αναφέρω είναι το Ισραήλ δεν χάνει ευκαιρία να καταφέρεται κατά του Ισραήλ με τρόπο αντισημιτικό το Ιράν. Η κατάσταση αυτή είναι αφόρητη. Δηλώνει δημόσια το Ιράν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη. Και το τέταρτο και τελευταίο είναι ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα πυρηνικά και τις κυρώσεις. Είναι ευαίσθητο αυτό το κεφάλαιο και ε, δεν υπάρχει ομοφωνία ε, στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ε, ε, βλέπει το, Ιράν να συνεχίζει απερίσπαστο τις προσπάθειες του για πρόθεση στο πυρηνικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να δούμε τι συστάσεις θα απευθύνουμε σχετικά στην υπάτη εκπρόσωπο. Τέλος, συνάδελφοι, προσβλέπω σε εντατική συνεργασία μαζί σας. Γνωρίζω ότι Πολλοί συνάδελφοι παρακολουθούν πολύ κοντά την κατάσταση στο Ιράν και θα συμπεριλάβω τα όσα μου πείτε στην έκθεση, ιδιαίτερα το ρόλο των θεσμικών οργάνων για να δώσουμε συστάσεις στο Συμβούλιο, την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Προς το παρόν το αφήνω εδώ, σταματώ εδώ και ε, περιμένω να ακούσω τις πρώτες σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και πρόεδρε. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοπά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Φυσικά κάνουμε αυτή τη στιγμή μια καταρχήν συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, περιμένοντας να δούμε το κείμενο, ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε με πιο συγκεκριμένες προτάσεις και σκέψεις. Το Ιράν ε, αποτελεί αντικείμενο μεγάλου προβληματισμού, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την διεθνή κοινότητα γιατί παραμένει μια ενδυνάμει απειλή. Και η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων επιβεβαίωσε την επί της αρχής ενότητα της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορά τη μη αποδοχή των πυρηνικών σχεδίων της Τεχεράνης. Πρέπει όμως να σκεφτούμε και να αξιολογήσουμε κατά πόσο αυτές οι νέες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, γιατί γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι μέχρι τώρα η πολιτική κυρώσεων απέναντι στο Ιράν δεν έχει αποδώσει, και κατά πόσο θα προστατεύσουμε τον απλό Ιρανικό λαό από τις κυρώσεις αυτές. Πώς δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε, αν μπορούμε, για έξυπνες κυρώσεις που πλήττουν πραγματικά αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι αξίζει να δούμε τη συνολική εικόνα. Δηλαδή, να διευρύνουμε τη συζήτηση για τα πυρηνικά στη Μέση Ανατολή συνολικά. Το Ισραήλ, για παράδειγμα, δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση για μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και εικάζεται ότι έχει ήδη στην κατοχή του πυρηνικά όπλα. Και γιατί όχι να επαναφέρουμε τη συζήτηση για μια ελεύθερη από πυρηνικά Μέση Ανατολή. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες σχετικά, και στην τελευταία διάσκεψη του ΟΗΕ, τον Μάη του 2010, για τη μη διάδοση, όπου το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων κάνει λόγο για την ανάγκη πρακτικών βημάτων, παροτρύνοντας τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη, να συγκαλέσουν το 2012 μια περιφερειακή συνδιάσκεψη για τη δημιουργία μιας Μέσης Ανατολής απαλλαγμένης από πυρηνικά και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής. Νομίζω είναι μια ιδέα που αξίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να συζητήσει. Τέλος, επειδή το έθιξε ήδη και ο εισηγητής και νομίζω είναι πολύ σοβαρό θέμα, είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, μέσα στη χώρα, η οποία πραγματικά είναι δραματική και εδώ ε, θα ήθελα απλώς να θέσω έναν προβληματισμό κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρει τρόπου στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, τρόπου στήριξης μιας κοινωνίας η οποία πραγματικά πλήττεται από το καθεστώς και έτσι από κάτω να δημιουργηθεί ένα κίνημα αλλαγής, από κάτω προς τα πάνω, στηρίζοντας την κοινωνία πολιτών, ενισχύοντας και ε, προωθώντας την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο Ιράν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Λόχμπιλερ που είναι και πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με το Ιράν. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ και κύριε Μπέλντερ για την εξήγηση πώς θα ε, διαρθρώσετε την έκθεσή σας. Συμφωνώ με τη βασική δομή. Θα ήθελα όμως να συστήσω το εξής. Το κεφάλαιο 3 που είπατε ότι είναι εξωτερικές σχέσεις και οι σχέσεις του Ιράν με την περιφέρεια και τους κινδύνους και τις ευκαιρίες θα παρακαλούσα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί τουλάχιστον στην περασμένη θητεία, συγγνώμη, πέρυσι διορθώνει ο Μιλήτρια, δεν ασχοληθήκαμε αρκετά εντατικά με αυτό το θέμα. Είχαμε ψηφίσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα πυρηνικά. Ε, όχι γι' αυτό και θα ήταν πολύ σημαντικό και συνεργασία με τις άλλες αντιπροσωπείες του Κοινοβούλιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορα think tanks, ομίλους προβληματισμού, να δούμε πώς ε, μπορεί να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική για το Ιράν που να εξετάζει και να ασχολείται με την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και ε, τι γίνεται στο Ιράκ, το Αφγανιστάν αλλά και πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους ε, να έχουμε μία μέση ατολή χωρίς πυρηνικά. Εδώ χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες και θα μπορούσαμε ενδεχομένως να προσθέσουμε και κάτι άλλο στο κεφάλαιο αυτό. για μια ευρωπαϊκή πολιτική για το Ιράν και για την εφαρμογή της θα πρέπει να υπάρχει επιτόπου αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να δούμε τα υπέρ και τα κατά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας τέτοια ε, ε, Αναφέρθηκε στην στην πολιτική κυρώσεων. Θα πρέπει να μελετήσουμε κατά πόσο έχουν αποτέλεσμα οι κυρώσεις που ήδη έχουν επιβληθεί με στόχο συγκεκριμένες ηγετικές ομάδες της ελίτ της χώρας. Αλλά θα πρέπει να αξιολογήσουμε μήπως πλήττεται από τις κυρώσεις αυτές και ο πληθυσμός και ο ευρύτερος πληθυσμός του Ιράν και τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Αυτό θα το συζητήσουμε μάλλον στο πολιτικό κεφάλαιο. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα είπατε ότι θα είναι πολύ μεγάλο αυτό το κεφάλαιο, όπως ε, και στα άλλα ψηφίσματα. Θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω κάτι ε, σημαντικό. Η κατάσταση του γυναικείου κινήματος να μας ε, προβληματίσει έχουν ε, ληφθεί πολλές πρωτοβουλίες και θα, υπάρξει μια, πρέπει να υπάρχει μια πολιτική κατά των διακρίσεων. Ευχαριστώ. Κύριος Πρέντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, να σας παρουσιάσω τη δική μας προοπτική. Και πώς βλέπουμε το θέμα από τη δική μας πλευρά. Πρώτα-πρώτα σας ευχαριστώ για την παρουσία σας κύριε Σιγητά. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράν είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Γιατί ε, εδώ δεν δράσαμε σωστά σε σχέση με τις ευθύνες που είχαμε αναλάβει βάσει της συνθήκης NDP. Και για το πρόγραμμα της ανάπτυξης πυρηνικών στο Ιράκ. Εδώ, όπως έχει υποθεί, η συνολική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχώς υποβαθμίζεται. Και μιλάμε εδώ για τα δικαιώματα των πολιτών και τι θεμελιώδει πολιτικέ ελευθερίε. Θα ήθελα να τονίσω τρία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα των πυρηνικών, των των πυρηνικών. Για το ΕΛΚ το τοσχέ αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σκέλος της προσέγγισης μας. Είναι σημαντικό το Ιράν να εκπληρώνει τις διεθνείς του υποχρεώσεις συγγνώμη, και να αναστείλει οποιαδήποτε πυρηνική δραστηριότητα. Το Ιράν έχει ήδη περιφρονήσει τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας και εφόσον δεν συμμορφώνεται, προφανώς θα συνεχίσει να εκτίθεται και να διακινδυνεύει διεθνείς κυρώσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τα μέτρα που προτείνονται στο ψήφισμα 1929 από τον Ιούνιο και όσο για τα μέτρα από, ευρωπαϊκή, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Η ιδέα αυτή είναι πολύ καλή, παρόλο που θα μπορούσαμε να έχουμε και διαπραγματεύσει για να εξεύρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση το Ιράν ε, βρίσκει πάντοτε τον καταλληλότερο τρόπο για να παρακάμπτει τα μέτρα και τις κυρώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δημοκρατικό πολίτευμα στο Ιράν, αυτό θα πρέπει να είναι ένα δεύτερο σκέλος της πολιτικής μας για το Ιράν και για το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 22 Οκτωβρίου για τη στήριξη της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις θα πρέπει να τονίσουμε τι γίνεται με την κοινότητα των Μπαχάη οι οποίοι ακόμη διώκονται και ο κύριος Μπούζεκ καταδίκασε τη στάση του Ιράν σε έναν από τους λόγους του. Θα πρέπει να μιλήσουμε επίσης για τους εξορίστους, οι οποίοι διώκονται ή είναι θύματα εκβιασμού από τις Ιρανικές αρχές. Για το ΕΛΚ τα ζητήματα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Το Ιράν διαρκώς παρεμβαίνει στα εσωτερικά των γειτονικών χωρών, όπως του Ιράκ, και στηρίζει τις τρομοκρατικές οργανώσεις που αποσταθεροποιηθούν το σύνολο της γεωγραφικής αυτής περιοχής. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που θέλω να αναφέρω. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Μουνής, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι λογική η παρουσίαση του εισηγητού ως προς το σκελετό της έκθεσής του. Τα μεγάλα κεφάλαια είναι ακριβώς αυτά, το πυρηνικό φαινόμενο, όπου η σοσιαλιστική ομάδα υποστηρίζει την προσέγγιση της διπλής οδού. Δηλαδή, να υποστηρίζουμε τις κυρώσεις με μεγάλη αυστηρότητα για την τήρησή τους, αλλά ταυτόχρονα να ε, Τίνουμε και μια χείρα συνεργασίας προς το Ιράν για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις, αν θέλει, για τα πυρηνικά. Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει βεβαίως να γίνει αναφορά σε αυτά στην έκθεση, ιδιαίτερα πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη και αδιάκριτη πρόσβαση του λαού στις τεχνολογίες ε, ε, πληροφορίες και να υποστηρίζονται ε, τα πολυφωνικά κινήματα αντιπολίτευσης. Χωρίς να μιλάμε για κάποια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη ή θρησκευτική κοινότητα. Υπάρχει το λεγόμενο πράσινο κίνημα ε, που είναι ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα και θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση. Και τέλος, ε, ο ρόλος του Ιράν στην περιοχή είναι πολύ σημαντικό. Είναι περιφερειακή δύναμη το Ιράν και έχει μεγάλη στρατηγική αξία και σίγουρα επιρροή στους γείτονές του. Αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε εμείς τώρα στο θέμα του Ισραήλ και την αντισημιτική θέση του Ιράν. Θα πρέπει να υπερβούμε αυτό το στοιχείο και να το, ξεπεράσουμε, δηλαδή να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, τις αραβικές χώρες, τις γειτονικές χώρες, να μην κολλήσουμε στο Ισραήλ. Και χώρες μουσουλμανικές κοινωνικά, όπως είναι η Τουρκία, αλλά ε, κοσμικές και όχι θεοκρατικές από πολιτικής πλευρά, να ξεφύγουμε από τον αντισημιτισμό και το Ισραήλ και να δούμε το ρόλο του Ιράν ευρύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σάρκε. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε και συνάδελφοι. Πολλά υπόθηκαν ήδη. Θα ήθελα λίγο να σταθώ, αν μου επιτρέπετε, στις κυρώσεις που είναι στην ημερήσια διάταξη και πάλι για το Ιράν και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη και να φροντίσει ε, τελικά να είναι ε, ένα παιχνίδι με αποτέλεσμα ουδέτερο και για τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα, zero sum. Θέλουμε να επικρατήσουν περισσότερες ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα ε, και να πιέσουμε το Ιράν προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και το ρόλο του εμπορίου, όχι μόνο στις κυρώσεις, γενικότερα, ως ε, σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας απέναντι στο Ιράν και να δούμε και τις ανεπιθύμητες ε, ενέργειες και επιδράσεις ε, στις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων. Υπάρχουν κάποιοι σκληροπυρηνικοί και συντηρητικοί όπως είναι η φρουρά της Επανάστασης σε περίπτωση κυρώσεων κερδίζουν σε επιρροή και αυξάνεται ο ρόλος τους. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Και ε, ο ΙΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ε, όταν θέλουν να επιβάλλουν νέες κυρώσεις μήπως ενισχύσουν ενδεχομένω κάποιες ομάδες που δεν θα επιθυμούν. Και επίσης στην εξαγωγή τεχνολογίας έχουν πάει πολλά πράγματα στραβά ε, και συχνά ε, αυτό το έχουν καταχραστεί ε, ολοκληρωτικά καθεστώτα, ε, το θέμα της τεχνολογίας, για να φακελώνουν, να παρακολουθούν το λαό και να στρέφουν αυτά τα εργαλεία της τεχνολογίας εις βάρος του λαού. Εντάξει η τεχνολογία, εντάξει το διαδίκτυο να έχει ελεύθερη πρόσταση ο λαός, αλλά όχι καταχρήσεις στα τεχνολογικά ζητήματα. Να δούμε τι γίνεται με τα μίντια και τις νέες μορφές μέσων επικοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία να υπάρξει και ένα άνοιγμα στο Ιράν προς τον έξω κόσμο για να λάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες, ας πούμε ε, εκπομπές φαρσί στην Ευρώπη. Και κάτι άλλο, πώς μπορούμε εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κοιτάξουμε το χρονισμό, το timing, πότε θα βγει αυτή η έκθεση, ε, ε, όχι κατόπιν ε, εορτής όταν θα έχουν ληφθεί οι διεθνείς αποφάσεις και να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με την Τουρκία που είναι μια χώρα πάρα πολύ σημαντική για την Τουρκία και σε σχέση με το Ιράν. Με τρόπο επικοδομητικό θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη χώρα αυτή για να προσέξουμε πάρα πολύ την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε ε, επί τσεχικής προεδρίας και λέγεται Shelters Cities. Για τους ακτιβιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων και εκπροσώπους αντιπολίτευσης να τους δώσουμε ενδεχομένως μια προσωρινή προστασία στην Ευρώπη. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ κάνει πολύ λίγα πράγματα η Ευρώπη, έχω την εντύπωση. Εάν εξετάσουμε κυρώσεις. Να δούμε τι σημαίνει αυτό και για την αντιπολίτευση και την πολιτική αντιπολίτευση και τι μπορούμε εμείς στην Ευρώπη να κάνουμε, τι μας αναλογεί ως μερίδιο ευθύνη. Έτσι, προς τα εκεί σκέφτεται η δική μας πολιτική ομάδα. Προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία, όπως είχαμε και στο παρελθόν, συναδέλφους από άλλες πολιτικές ομάδες, για το Ιράν. Ευχαριστώ. Κυρία Λούζινγκ, παρακαλώ. Για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρώτα. Όποιο έχει συμφέρον και ενδιαφέρεται για εκδημοκρατισμό του Ιράν θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε ε, να ε, αποσοβηθεί ένταση σε διεθνές επίπεδο. Οποιαδήποτε κλιμάκωση ε, απειλεί με μείωση της δημοκρατίας στο εσωτερικό της χώρας και μείωση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Η μέχρι τώρα πολιτική της σύγκρουσης και της απομόνωσης του Ιράν από τη Δύση οδήγησε σε πραγματικό αδιέξοδο. Η συνέχιση τώρα με νέα μέτρα, με νέες κυρώσεις, αφού αποδείχθηκαν οι προηγούμενες άχρηστες, και αν έχουμε τώρα επίθεση στο Ιράν, παρά, βιάζοντας το διεθνές δίκαιο, αυτό θα είναι εις βάρος όλων των πάντων. Ερώτηση. Τι δυνατότητες υπάρχουν, τι συμφέρον υπάρχουν εκατέρωθεν, να βρούμε στόχους ρεαλιστικούς και να τους εφαρμόσουμε στη διαπραγμάτευση. Το 2009 έγιναν δημοσκοπήσεις στο Ιράν και 72% του πληθυσμού ε, είναι υπέρ των επιθεωρήσεων και έτσι εγγύσεις να μην υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Αν η τεχνολογική βοήθεια δοθεί από άλλα κράτη ε, και βεβαίως με ευρύτατο διεθνή έλεγχο. Αυτή την προοπτική θα πρέπει κατά την άποψή μου να τη λάβουμε υπόψη μας. Και Μέχρι τώρα, ε, όταν κάποιος θέλει να αναπτύξει πυρηνικά, θεωρεί ότι απειλείται από κάπου. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε εμεί πώς απαντούμε σε αυτό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε να δώσουν αξιόπιστες εγγυήσει ότι δεν θα επιτεθούν στο Ιράν. Και ποιο ρόλο μπορεί να παίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όλο ακούμε για σενάρια απειλής του Ιράν. Μα αυτά τα σενάρια απειλής ε, έχουν πολύ διαφορετική αξιολόγηση και αυτό δεν έχει να κάνει με αριστερά, δεξιά, πολιτική και τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να δούμε και τι λέει η CIA. Και αυτοί πολύ διαφορετικά αξιολογούν την απειλή. Ο Ντένις Πλέερ επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών είπε το 2010 στην Αμερική ότι θεωρούμε ακόμα ότι το Ιράν διατηρεί ανοιχτή αυτή τη δυνατότητα και το ενδεχόμενο και δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση θα αποφασίσει. Και συνεχίζει. Παραμένουμε στην αντίληψη ότι η ανάλυση κόστους ωφέλειας θα ε, μας οδηγήσει στην απόφαση Μάλλον θα, οδηγήσει το Ιράν ε, στην απόφαση του προς τη μία την άλλη κατεύθυνση και το περιβάλλον του Bill Clinton, ο Τζόζεφ Νάι, καθηγητής στο Χάρβαρτ, είπε θα πρέπει να έχουμε στόχο να πείσουμε την Τεχεράνη να ακολουθεί στο δρόμο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν πυρηνική ενέργεια, μπορούν να ε, φτιάξουν πυρηνική ατομική βόμβα, αλλά αποφάσισαν να μην το πράξουν. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η προοπτική και αυτός ο δρόμος στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το Ιράν και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς αυτή την ε, πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάντλενερ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία λόγια όλα αυτά. Τα ε, ε, βρίσκουμε πολύ ωραία και τα συμφωνούμε. Καλό θα ήταν το Ιράν να είναι ελληνικό, αλλά έχουμε που χτίσει. Είναι ένα βαρβαρικό, ισλαμικό, τρομοκρατικό καθεστώς που κάνει εγκλήματα κατά της ίδιας κυβέρνησης που κρεμάει πολιτικούς αντιπάλους. Ο Αχμαντή Τζάν έχει αίμα στα χέρια του και θα πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρο ότι για μας είναι απαράδεκτο αυτό το καθεστώς ε, τρόμου να συνεχίσει. Και με χλιαρά κείμενα για κατευνασμό, appeasement, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα πούμε σκληρά, γιατί είναι σκληρά αυτά που γίνονται. Τα είπε και ο εισηγητή με ισχυρή γλώσσα και ισχυρές επιλογές. Να μην είμαστε χλιαροί. Και ποιος είναι ο ρόλος του συμμάχου μας. Η Τουρκία ε, κάνει περίεργη πολιτική για το Ιράν και υπονομεύει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία απομόνωσης του Ιράν. Ο Ερτογάν λέει, ε, αποκαλεί μεγάλο του φίλο τον Αχματίν Νετζάν. Αυτό δεν θα πρέπει να το θεωρούμε καλό όταν διαπραγματευόμαστε με την Τουρκία. Απαράδεκτο είναι. Και έχει και πυρηνικές φιλοδοξίες ο Αχματίνετζάν και τον βοηθάει η Τουρκία. Μα αυτά είναι άλογα πράγματα, άφρονα. Θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία στην απομόνωση του Αχματίνετζάν. Είναι απαράδεκτα αυτά που κάνει η Τουρκία και να τις τα πούμε έξω από τα δόντια. Και ο σύμμαχός μας η Κίνα και ο εμπορικός μας εταίρος πάντα διστάζει να επιβάλλει κυρώσεις και αυτό θα πρέπει να το καταγγείλουμε. Έχουμε μεγάλους δεσμούς με την Κίνα, συγγνώμη να τους ε, εξηγούμε και σε εκείνου ε, ποια είναι η βαρβαρότητα. Και η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να απομονωθεί. Τονίζω το ρόλο της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης, τα είπαν κι άλλοι. Ήδη έχουμε πολλούς πρόσφυγες στην Ευρώπη που έχουν και πολλές επαφές ε, και υποστηρίζω αυτό. Ο ρόλος κυρίας Άστον Δεν κάνει τίποτα. Τι να πάει να κάνει εκεί η κυρία Άστον. Ε, λέει και αυτή κάτι χλιαρά με τους ηγέτες εκεί. Δεν έχει νόημα. μην είμαστε αφελείς, σε πάση περιπτώσει. Το Ισραήλ ευτυχώς έχει μεγάλη θέση και σαφή στο αντίστοιχο κεφάλαιο του εισηγητού και το υποστηρίζουμε πάρα πολύ γιατί ε, είναι τρομακτική και η γλώσσα ακόμα που χρησιμοποιεί το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ και θα πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα και οξύτατα οι προληπτικές ε, ε, επιθέσεις, preemptive strikes, δεν το θεωρεί απειλή αυτό τζατ. Δεν λέμε ότι θα πρέπει να γίνει, αλλά αν χρειαστεί τι να κάνουμε. Είναι τρελός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να ε, αποκτήσει πυρηνικά όπλα, πυράβλους που να τους στρέψει κατά του Ισραήλ. Λοιπόν, όχι πολιτική κατεγνασμού, κανένα appeasement, ε, πλήρης απομόνωση. Όχι να το συζητάμε με τον Αχματίνετζάν, να τον συλλάβουμε. Θα παρακαλούσα τον εισηγητή να σκεφτεί και αυτή τη γραμμή να τη βάλει στην έκθεσή του. Thank you very much. Now, uh, Mrs. Gomes, please. Η κυρία Γκόμες. Το Ιράν είναι σαν ένα από τα πολλά καθεστώτα που δεν μας αρέσουν και από τους ανθρώπους που δεν συμπαθούμε, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, πρέπει να τα καταφέρουμε και να μην αποφύγουμε και τις αποτρόπες συνέπειες της ύπαρξής τους. Προφανώς δεν συμφωνώ με μια προληπτική επίθεση κατά του Ιράν. Οποιαδήποτε τέτοια ιδέα δεν με βρίσκει σύμφωνη. Δεν πρόκειται να δουλέψει κάτι τέτοιο. Δεν είναι συνετό και οι συνέπειε ήταν τραγικέ για όλη την ανθρωπότητα και για την περιοχή και για το Ισραήλ. Πρώτο πρώτο. Πιστεύω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, δραστικό ρόλο να διαδραματίσουν. Και θα πρέπει να τις παρακολουθούμε εδώ. Είναι η δύναμη που έχουν παρεμποδίσει όσους θα ήθελαν να εξαπολύσουν μια προληπτική επίθεση και ξέρουμε ότι τέτοιες φωνές ακούστηκαν στο Ισραήλ. Έπειτα, το θέμα είναι πώς θα συνεργαστούμε με το Ιράν και τι μπορούμε να απαιτήσουμε από το Ιράν. Αυτό που πρέπει να απαιτήσουμε από το Ιράν είναι να μην συνεισφέρει στην εξάπλωση των πυρηνικών, τη διάδοση μάλλον των πυρηνικών. Και εγώ δεν πιστεύω ότι το Ιράν δεν έχει κανένα πυρηνικό στρατιωτικό πρόγραμμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, Ιδάλω, γιατί σε άλλη περίπτωση μόνο το Ιράν δεν ε, θα είχε παραβλέψει τελείω την IAA. Δεν θα είχε λοιπόν να αποκρύψει τίποτα από την IAA. και ίσως να αποτελέσει παράδειγμα το Ιράν αν έχει πυρηνικό στρατιωτικό πρόγραμμα και για άλλε δυνάμεις στην περιοχή ώστε να ακολουθήσουν πυρηνικού στόχους. Για αραβικές δυνάμεις συγκεκριμένα και αυτό αποτελεί απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ακόμη λοιπόν και αν το Ιράν ισχυρίζεται ότι δεν χρησιμοποιεί τα πυρηνικά για στρατιωτικού σκοπού, με τη στάση που τώρα τηρεί, πραγματικά είναι είναι ανεύθυνο στη στάση του και, δείχνει ότι και μπορεί να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επίσης πιστεύω ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωση εδώ πρέπει να είναι απόλυτα συνεπής. Πιστεύω ότι η διεθνή κοινότητα δεν έχει πετύχει στη δράση της και στο διάλογο με, με το Ιράν λόγω ασυνεπιών επί κυβέρνηση Bush οι υπεύθυνοι τη Αμερικανική κυβέρνηση δεν δέχονταν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με του ε, συνομιλητέ του από το Ιράν. Ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει με την κυβέρνηση Ομπάμα βέβαια και έχει αλλάξει και το μήνυμα που έχει αποσταλεί προ το Ιράν. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και πολύ σταθεροί προ τι κυρώσει όπω αυτέ που πρόβλεψε το Συμβούλιο Ασφαλεία το ΙΕ τον περασμένο Ιούνιο. Και ω προ αυτό να πω ότι βεβαίω οι κυρώσει δεν αποκλείουν το διάλογο με το Ιράν, όμως ο διάλογος θα πρέπει να έχει προγραμματιστεί προσεκτικά. Ε, ο Ιρανός Υπουργός αυτή τη στιγμή περιοδεύει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και εγώ δεν βλέπω από, αυτούς να υπάρχει, από αυτές τις συζητήσεις να υπάρχει κανένα όφελος. Μόνο για να σταματήσει κάπως αυτό το κλίμα πολιτικού και διπλωματικού αποκλεισμού του Ιράν που έχει δημιουργηθεί με τις πρόσφατες κυρώσει. Πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ είναι σημαντική η διάδοση των ειρηνικών να μην δώσει την εντύπωση σε όλους ούτε στο Ιρανικό καθεστώς ούτε στον Ιρανικό λαό που πολεμάει για την ελευθερία της δημοκρατίας και τι βασικέ ελευθερίε και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Να μην δώσει λοιπόν την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ξεπουλήσει όσου αγωνίζονται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν για να βρει μια λύση για τον φάκελο των πυρηνικών. Και οι δύο επιλογές αυτές είναι εξίσου σημαντικές και οι δύο κατευθύνσεις, αλλά καμία δεν είναι ανταλλάξιμη σε σχέση με την άλλη. Ε, δεν μπορεί να οδηγήσει σε κατάληψη της άλλης. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τι δύο κατευθύνσει παράλληλα και σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και τι ΗΠΑ. Άκουσα πολλού ε, υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο, που εργάζονται στο Ιράν, ιδίω μέσα από μια κρόαση που οργάνωσε η πολιτική μου ομάδα. Άκουσα τι εμπειρίε του και ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε και άλλε τέτοιε ευκαιρίε για να εξερευνήσουμε τι δρόμοι υπάρχουν και τι ελεύθερα μέσα μαζική επικοινωνία θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον Ιρανικό λαό τα πολιταρχικά, αυταρχικά καθεστώτα, τα διδακτορικά καθεστώτα, στόχο έχουν να παρεμποδίσουν την ελεύθερη ροή πληροφοριών προς το λαό. Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει μια κοινωνία ιδιαίτερα μορφωμένη, πολύ προηγμένη στο Ιράν, αποζητά την πρόσβαση στα νέα μέσα επικοινωνίας, στις νέες τεχνολογίες, αλλά είναι και θύμα της τεχνολογίας ε, ελέγχου της πληροφορίας, του τζάμιν. Θα πρέπει λοιπόν να προταθούν δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις, να προστατεύσουμε την κοινωνία των πολιτών στο Ιράν και αποτρέποντας τις απόπειρες jamming, δηλαδή τις, ε, του ελέγχου της πληροφορίας που προσφέρονται στους πολίτες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις τους. Τα σημείωνα αλλά πολύ σοβαρά. Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών θα μελετήσω και θα γράψω και ελπίζω το Σεπτέμβριο να φέρω γρήγορα ένα κείμενο. Θα τολμούσα να διαπιστώσω ότι τα τέσσερα κεφάλαια που ανέφερα εσωτερική πολιτική κατάσταση, ανθρώπινα δικαιώματα, εξωτερικές περιφερειακές σχέσεις και τα πυρηνικά είναι κάτι που ενδιαφέρει όλα τα μέρη που μίλησαν και τόνισαν όλοι ότι πραγματικά θα πρέπει να ασχοληθούμε ε, μεθοδικά και με τα τέσσερα θέματα, να δούμε ποιες είναι οι θέσεις της Επιτροπής Εξωτερικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο και το για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε σαφή θέση τελικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε λόγος πολλές φορές και σε λεπτομέρειες και από μια Ισπανίδα συνάδελφο που είπε να μην μας ενδιαφέρει μόνο ε, καμιά αλφαβήτα θρησκευτική μειονότητα ή ένα κράτος. Μα εμείς θέλουμε να δούμε τι κάνει το Ιράν, το καθεστώς του Ιράν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και πώς αυτό προάγει ή εμποδίζει τις εύρυθμες σχέσεις του Ιράν με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κόσμο ολόκληρο ή αν αποστεθεροποιεί. Γι' αυτό το αναφέρω. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις εθνικές μειονότητες και τις σκεφτικές στον πληθυντικό, όχι για μία. Και η κυρία Γκόμες είπε θα πρέπει να είναι μια κοινωνία όπου μπορεί ο λαός να αναπνέει ελεύθερα και η ελευθεροτυπία και ε, σας επαναλαμβάνω για τον έντυπο τύπο και για τον ηλεκτρονικό. Τέλος, Πρόεδρε, και ε, σύντομα άκουσα πολλά που θεωρώ χρήσιμα, τα σημείωσα, θα τα συμπεριλάβω στην έκθεσή μου και να είναι βέβαιοι συνάδελφοι ότι θα κάνω αντικειμενική έκθεση με ειλικρίνεια, θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα και θα δούμε και το θέμα των κυρώσεων. Η πολιτική κυρώσεων μπορεί να γίνει με πιο ευφύ τρόπο, με καλύτερο τρόπο και επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε πότε θα κατατηθεί η έκθεση. Αν έχω ενημερωθεί καλά το Συμβούλιο στις 16, 26 μάλλον ε, Ιουλίου θα αποφασίσει ε, εάν θα επέλθουν νέες κυρώσεις ε, δηλαδή να συνοδεύουν ε, τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές. Θα μπορούμε και αυτό να τα συμπεριλάβουμε λοιπόν στην έκθεσή μας για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, σε γενική ανάλυση, ευχαριστώ πολύ. Ήξερα ότι είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και η προσήλυξη του Κοινοβουλίου για το Ιράν. Το διαπίστωσα και πάλι και Προσβλέπω στην επόμενη φάση τώρα σε άλλες συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε την έκθεση μετά το καλοκαίρι. Και εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, γιατί τις έχουμε όλοι ανάγκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι που ξέχασα να σας πω ότι το, όριο ομιλίας για κάθε ομιλητή ήταν 20 λεπτά σε αυτή τη συζήτηση. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Το σεβαστήκατε όλοι πάντως έτσι κι αλλιώς. Να ευχαριστήσω και εσάς και τους διερμηνείς. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους Ισπανούς και τους ε, Ολλανδούς ε, για την εξαιρετική εκδήλωση και σας ευχαριστούμε, ε, σας ε, ευχόμαστε καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι.